Präsident! Darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Καθίστε παρακαλώ. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße σας καλωσορίζω και έρχεται η συνεδρίαση. Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υπομορφή ε, δήλωση του καγκελαρίου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Αυστρίας, τον κύριο Βέρνερ Φάιμαν, τον οποίο ορίζω. Καλώς ήρθατε κύριε καγκελάριο. Κυρίες και κύριοι, είδα κατά τη διάρκεια... Βλέπω εδώ πέρα πώς εκπροσωπείται η κυβέρνηση της Ισπανίας από τον ε, επί των ετών μου κύριο Ινίγκο Μέντες, Μέντες Δεβίγκο στα έδρανα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Κύριε Καγκελάρια, σας ευχαριστώ για το ότι δεχτήκατε την ε, πρόσκλησή μου να έρθετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να μιλήσετε με τους ε, βουλευτές μας για το πώς βλέπετε εσείς το μέλλον της Ευρώπης. Οπωσδήποτε το φέτος, το 2013, βρισκόμαστε σε μια αποφασιστική φάση της ε, πολιτικής ε, στην Ευρώπη και χωρίς καμία αμφιβολία η συνοχή των λαών και των κρατών στην ε, κοινότητά μας, μια κοινότητα κρατών και εθνών, έχει αποφασιστική σημασία για το πώς θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη το μέλλον, το οικονομικό, το οικολογικό και το νομισματικό και νομίζω πως πηγαίνουμε προς μια κατεύθυνση την οποία εγώ και εσείς φαντάζομαι πριν μερικά χρόνια δεν θα μπορούσατε να την είχατε φανταστεί. Η συζήτηση λοιπόν του Κοινοβουλίου μας με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με εσάς δηλαδή ως μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ταυτόχρονα επικεφαλής κυβέρνησης μιας κυρίαρχης χώρας έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό, επαναλαμβάνω, πως σας ευχαριστώ που ήρθατε ως εδώ για να συζητήσουμε μαζί. Και θα ευχόμουν περισσότεροι συναδελφοί σας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ε, έρχονταν ως εδώ και να έκαναν διάλογο με τους ε, ερετούς εκπροσώπους των λαών της ε, ευρωπαϊκής ε, κυβέρνησης από το να κάνουν δηλώσεις ε, ως εκπρόσωποι μιας χώρας στο έδαφος μιας άλλης χώρας. Και νομίζω πως θα συμφωνήσει μαζί μου και η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών. Τον λόγο τώρα έχει ο καγκελάριος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Αυστρίας, ο κύριος Φάιμαν. Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, χαίρομαι για το ότι βρήκατε το χρόνο να έρθετε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, για μένα είναι μια ιδιαίτερη τιμή να παρευρίσκομαι εδώ και να